La séance est reprise. Συνεχίζεται η συνεδρίαση και στην ημερήσια διάταξη έχουμε ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία είναι για την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Αγγελιλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκαταβολικές πληρωμές ε, στο πλαίσιο του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. 17 μάλλον. Ε, η η κυρία Πατρίτσια Σουλή. Amendement numéro 1, qui est pour. Ah, peut-être devons-nous faire un... Ε, να κάνουμε έναν έλεγχο πριν ε, ξεκινήσουμε για να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Δοκιμάστε παρακαλώ για να δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί. Πέρασες της ψηφοφορίας. για την ε, έκθεση της κυρίας Σιλίνη. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου Ολοι Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορία. Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Σουλίνη έκθεση του κυρίου Βιώτη, γνωμοδότηση. Σχέδιο γνωμοδότηση για την αντιμετώπιση των μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, ο ρόλο τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 και 7 που είναι οι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται μάλλον, τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, επαλήθευση με ηλεκτρονική ψήφο. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ, κατά, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 14 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Η 17 που σύρθηκε 18 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 22 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, επαλήθευση. Πέρυσι Απορρίπτεται. 15 κατά 11 υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Βιώτη. Και τώρα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου μας Νοβάκοφ για την εφαρμογή του έρασμος ΣΥΝ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Α, ε, Απορρίπτεται 13 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας όλοι. Ποιοι είναι υπέρ, ξαναρχίζουμε. Ευχαριστώ, κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 11 με 16. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 11-16. Τροπολογία 5 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ Α, για την 5 που είναι συμβατή με την 4 ποιοι είναι υπέρ της 5 λέει ο πρόεδρος κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλά να ελέγξουμε Πέρας. Απορρίπτεται 13, 14. Ε, Τροπολογία 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. πέρας εγκρίνεται 15-13 τροπολογία 8 κατά αποχές να ελέγξουμε και εδώ πέρας απορρίπτεται 13-15 τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά να ελέγξουμε πέρας εγκρίνεται 15-13 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 14 με 9. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά να ελέγξουμε πέρας Απορρίπτεται 12 με 17. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 10-18. Σας παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 αν ελέγξουμε καλά ελέγχουμε την 32 πέρας εγκρίνεται με συγχωρείτε 33 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Με συγχωρείτε. Α, α υπάρχει και προφορική τροπολογία του συγκεκριτή. Μάλιστα. Με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και στο σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά Πέρας. Εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Structural Πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η έκθεση Olbricht. Λοιπόν, θα σας πρότεινα να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες που στοχεύουν να απαλείψουν τα μέτρα αυτά. Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Όχι. Ωραία. Θα ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 12 καταρχάς. Υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν αυτή η κοινή ψηφοφορία για τις τροπολογίες απόρριψης. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή η κοινή ψηφοφορία. Και πάμε στην τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 89, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται, 15-12. Τροπολογία 92 και 93 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 αποσύρεται, το ίδιο και 100, Η 101 και 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104-105 ε, ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 106-107 <coughs> υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 109-10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 11-12 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 όμως η 117 ήταν τα, με την 116. Άρα έχουν απορριφθεί και οι δύο. 120-121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 126 αποσύρεται. 129-130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 134-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η τροπολογία 5 που θα ψηφιστεί από κοινού με την τροπολογία 7 υπέρ κατά εγκρίνονται. 140 υπέρ 140 υπέρ λοιπόν κατά αποχές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 15-11. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146-7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 ε, ψηφίστηκε με την 5 unblock. 158 υπέρ. Α, κατά απίπτη. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ όχι κατέπεσε καλύπτεται από την 8 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 και 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 205 αποσύρεται 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 13 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 και 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, α, κατέπεσε. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 56 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. «58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται» και 59 μαζί. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, απο, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατέπεσε, γιατί καλύπτεται από την 4, 67 υπέρ, όχι, κατέπεσε και αυτή. Συμβατή με την 4. Ή μάλλον θα την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά για την 67. 67 συμβατεί με την 4. Υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Ψηφίζουμε. Όχι. Γιατί κατέπεσε η 68. Επομένως 69 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Πέραση ψηφοφορία Απορρίπτεται. 11 ψήφοι. υπέρ, 17 κατά. Στο σύνολο του κειμένου, η ηλεκτρονικά. Ε, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στον κύριο Όλμπριχτ. Γνωμοδότηση της κυρίας Χολμάιερ ε, αναβάλλεται, επομένως θα ψηφίσουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση της κυρίας ε, Γκαρδιά Θαμπάλ για το, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 11 ψήφοι υπέρ, 17 κατά δεύτερον τμήμα υπέρ, κατά εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται 15 ψήφι υπέρ, 13 κατά. 12 υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της κυρίας Γκαρδία Θαμπάλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Πέραση ψηφοφορίας, απορρίπτεται, ναι, αλλά σηκώντε τα χέρια σας παρακαλώ. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, δεκτή, 16 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ 14 κατά 17 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 17 ψήφοι κατά, 11 υπέρ. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Καρδία Θαμπάλ. Ε, de Econ, la commission au fond, je ne sais pas si vous voulez le mentionner ou pas. Pour Econ. Je ne sais pas. La parole est maintenant à Rose Emmanuel Fernandez pour deux transferts. Να δώσουμε το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες για δύο μεταφορές πιστώσεων του τρέχοντος έτους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο μεταφορές λοιπόν. Το 32, 18 εκατομμύρια 200.000 ευρώ υποχρεώσεις και 2 εκατομμύρια 388.544 ευρώ πληρωμές. Αφορά διάφορες διοικητικές γραμμές διαφόρων ε, εκτελεστικών οργανισμών και δραστηριότητες επικοινωνίες για γραμμές λειτουργίας του προγράμματος COSME και προτείνω να το εγκρίνουμε. Και μετά έχουμε το 33, τη μεταφορά 33, 33 εκατομμύρια πληρωμές λόγω κάποιων καθυστερήσεων πληρωμών προς το έρασμο ΣΥΝ που σημειώσαμε μετά την γενική μεταφορά και όπου υπάρχει μεγάλη κατανάλωση πιστώσεων πληρωμών προτείνω να εγκριθεί και αυτή η μεταφορά πιστώσεων. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Για περαιτέρω διευκρινήσει. Ηλεκτρονικά λοιπόν παρακαλώ. Για τη μεταφορά πιστώσεων 32. Ε, ο εισηγητής ε, είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ και 2 κατά για την τροπολογία 33 και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ 2 κατά Είμαστε πάντα στον προπολογισμό του τρέχοντος έτους για τα άλλα τμήματα, το λόγο έχει ο Ζεράρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε 16 προτάσεις μεταφορών πιστώσεων. Μεταξύ τους οι 14 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν, αλλά υπάρχουν δύο επί των οποίων θα επανέλθω, όπου θα πρέπει να ψηφίσουμε. Μία πρώτη μεταφορά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η nf 2 του 2016, δεν δημιουργεί προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Κατόπιν έχουμε το enf 16 Έτοιμα μεταφοράς πιστώσεων του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή επίσης δεν θεωρώ ότι δημιουργούν προβλήματα. Το ελεκτικό συνέδριο έχει πέντε αιτήματα μεταφορών, είναι μικρά ποσά, κατά τη γνώμη μου επίσης δεν αποτελούν πρόβλημα. Η Επιτροπή Περιφερειών επίσης ε, ζητά πέντε μεταφορές πιστώσεων, δεν υπάρχουν προβλήματα επ' αυτών, αλλά θα επανέλθω θα επανέλθω σε αυτό που λέγεται DOSE 2016 για την ε, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τρία αιτήματα μεταφορών. Τα δύο δεν ε, είναι προβληματικά, αλλά θα επανέλθω επί του ε, ε, σε 1-2016. Αν συμφωνούν λοιπόν οι συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι 14 πρώτες μεταφορές δεν δημιουργούν πρόβλημα και μπορούν να εγκριθούν. Ο κύριος Μακά. Θα ήθελα να πω ότι εγώ στηρίζω την πρόταση του εισηγητή. Ε, θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξής. Αν δούμε λιγάκι την Επιτροπή των Περιφερειών, διαπιστώνουμε ότι κάθε χρόνο ε, κατά 5% η διερμηνία ανατίθεται κατά 15 περίπου περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το ίδιο διαπιστώνεται και για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι κάθε χρόνο απολύονται οι μόνιμοι υπάλληλοι 1% το χρόνο και αντικαθίσταται στη δουλειά τους από ελεύθερους συνεργάτες, freelance. Η Κομισιόν πρέπει να το δει και αυτό. Δηλαδή τι κάνουμε τελικά, υποτίθεται ε, κάνουμε κάποια εξοικονόμηση, απολύουμε τους υπαλλήλου και μετά τους ξαναπροσλαμβάνουμε ως ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εξοικονόμηση κονδυλίων. Πρόεδρος. Έτσι λοιπόν ε, δίνουμε την εντύπωση ότι μειώνουμε τις δαπάνες για το προσωπικό. Είναι μια δογματική προσέγγιση, αλλά ίσως να μας κοστίσει περισσότερο γιατί κατόπιν μετά πρέπει να προσλάβουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Και ό,τι δεν πληρώνουμε ως μισθούς, το πληρώνουμε ως παροχή υπηρεσιών. Ο πρόεδρος. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος Μπανκά. Είναι η άμεση επίπτωση της μείωσης 5% του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιες υπηρεσίες ε, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με υπαλλήλου και πληρώνουν περισσότερα για παροχή υπηρεσιών. Εγώ θα πει ήταν ηλίθια αυτή η πολιτική της μείωσης του προσωπικού. Πρόεδρος, λοιπόν, έχουμε τα δύο αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων για την Οικονομική και Κοινωνική ε, Επιτροπή. Είναι η μεταφορά 2S1 2016 και όσον αφορά την Επιτροπή Περιφερειών είναι, είναι η ίδια ακριβώς ε, ε, ε, αναφορά. Είναι σχετικά σημαντικές 1.274.000 και 935.800 ευρώ για την Επιτροπή Περιφερειών. Περί πρόκειται. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Περιφερειών και ε, ε, ε, έχει την έδρα της σε κτίρια στις Βρυξέλλες. Εδώ προτείνει να μεταφορθούν αυτές οι πιστώσεις, δεν επανέρχομαι στις τεχνικές λεπτομέρειες, για να κάνει το εξή. Θα μπορούσε να πληρώσει με βάση τις πιστώσεις του 16 και όχι τις πιστώσεις του 17 το κόστος της εμφυτευτικής μίσθωσης για το 17. Είναι θέμα του ετήσιου χαρακτήρα του προπολογισμού. Άρα αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αλλά για ορισμένου λόγους θεωρώ ότι μπορούμε να εγκρίνουμε. Πρώτον, διότι έχουμε εγκρίνει όλες τις μεταφορές για τον προπολογισμό του 2016, γιατί ήταν η επίσημη πρόταση της Επιτροπής και το δεχθήκαμε για το σύνολο των θεσμικών οργάνων. Δεύτερον, αν δεν αποδεχθούμε αυτή τη μεταφορά πιστώσεων, ούτως ή άλλως κάποιες πιστώσεις θα ακυρωθούν και που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση, για παράδειγμα, για λόγους ασφαλείας ε, του χολ της εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναβληθούν αυτές οι εργασίες και θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πιστώσεις για τον επόμενο προπολογισμό του 2017. Για αυτούς τους λόγους. Και επειδή δηλαδή για το σύνολο των ε, θεσμικών οργάνων όταν εγκρίναμε το σχέδιο προπολογισμού του 2016, το εγκρίναμε λοιπόν ως προσέγγιση για όλα τα όργανα, και επειδή πρέπει αυτές οι εργασίες για βελτίωση της ασφάλειας να γίνουν τάχιστα, θεωρώ ότι έχει σημασία να εγκρίνουμε αυτές τις δύο προτάσεις μεταφοράς πιστώσεων. Ευχαριστώ κυρία Χολμάια. Ήθελα να μιλήσει από αυτού. Ε, προηγουμένως Ε, ήθελα να μιλήσω λιγάκι για το θέμα αυτό τη ε, εξωτερικού συνεργάτες. Κοιτάξτε, ω Κοινοβούλιο έχουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, στην υπηρεσία της μετάφρασης και της ε, διερμηνίας κάναμε εξοικονόμηση πολύ μεγάλη σε προσωπικό. Βεβαίως, ε, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ότι θα πρέπει να μιλάμε για οργανόγραμμα αλλά όχι για τα οικονομικά στοιχεία. Και αυτό βέβαια ως κοινοβούλιο μας επλήξε. Κάναμε κάποιες εξοικονομήσεις. Αλλά αυτό δεν βοήθησε. Σωστό λέω, Πρόεδρε. Α, και ο κύριο Ζούμπι, Παρακαλώ. Όχι, α, καλά. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά και μαζί, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτές τις δύο μεταφορές. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις δύο μεταφορές που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Πέρας εγκρίνονται 23 ψήφοι υπέρ 2 κατά Κυρία Χολμάια δεν υπάρχει κανένα αίτημα για ψηφοφορία επί των ακινήτων Νομίζω ότι επί των 14 αυτών έχουμε ήδη εκφραστεί έτσι, δεν είναι. Δεν υπήρχε αντίρρηση. Ωραία. Θεωρούμε ότι 14 άλλες μεταφορές πιστώσεων έχουν ήδη εγκριθεί. Οπότε, λίγη ψηφοφορία. Οπότε, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Χολμάια για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ λοιπόν πρόκειται για μια περίπτωση η οποία ε, παρουσιάστηκε μέσω τηλεόραση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κυρίως πρόκειται για την περιοχή Ρούταλ Ιν, για την περιοχή της Κάτω Βαβαρίας ε, στη Γερμανία. Το Μάιο και Ιούνιο του 2016 αυτή η περιοχή επλήγει από πλημμύρες. Πέθαναν 7 άνθρωποι, 47.000 άνθρωποι ε, υπέστησαν ζημιές ε, και για να το πω έτσι και πάρα πολύ απλά μέσα σε δέκα μόνο λεπτά μια ολόκληρη πόλη βρέθηκε κάτω από το νερό και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν είτε να ανέβουν στον πρώτο όροφο, αν υπήρχαν ακόμα τα σπίτια τους, αν είχαν παρασυρθεί από τα νερά, προσπάθησαν να βρουν κάποια λύση. Κάποιοι όμως δεν τα κατάφεραν, ε, πάνω από 2.000 άνθρωποι κατέστησαν άστεγοι. Και η πόλη που επλήγει κυρίως ήταν η πόλη Ζίμπαχ Αμ Ιν. διακόπτη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ε, όσοι φεύγουν, σύντομα. Τώρα, το ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε στο τα λιγότερα εκεί στην περιοχή είναι 1,26 δις, πάνω από 3% του ε, εθνικού προϊόντος της κάτω Βαβαρίας. Άρα δηλαδή ξεπερνάει κατά 1,5 το περιφερειακό ΑΕΠ και Εκεί ορίζεται επίσης και η περιφερειακή καταστροφή όπου μιλάμε για 2,5 από 1,6 δις, αυτό το ποσό επιστρέφεται, δηλαδή καταλήγουμε σε 450 τόσες χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ε, είναι η συνηθισμένη, δηλαδή η Κομισιόν εξέτασε όλα τα στοιχεία και ως εκ τούτου ε, δεν υπάρχει τίποτα το φοβερό για να πούμε παρά μόνο το ότι ε, θα πέρασε ακόμα αρκετός καιρός μέχρι η πόλη αυτή η Ζήμπαχ να μπορέσει να λάβει τη μορφή που είχε και κατά το παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε Χολμάλη ο Πρόεδρος. Όλοι θυμόμαστε πόσο σοβαρή ήταν αυτή η καταστροφή. Οπότε, θέλει κανείς το λόγο. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ε, παρουσίαση, κυρία Χολμάια. Ίσως να υπάρξουν τροπολογίες που θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι αύριο 10 το πρωί. Η προφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν έχω, έχω καθορίσει όμως, δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία της, ούτε η ημερομηνία συζήτηση στην Ολομέλεια. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες που θα αναφερθεί σε τρεις διορθωτικούς προϋπολογισμούς για το 2016. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω αναφερθεί επανειλημμένο στο θέμα αυτό στην Επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε το τμήμα 5, είναι ένα τμήμα το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Είναι απλώς ε, μια αντιστάθμιση από την ε, εφαρμογή μιας απόφασης του 2014 για τους ίδιους πόρους και εδώ προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά το ε, Ταμείο Λελεγγύης για τη Γερμανία ε, για να βοηθήσουμε για τις πλημμύρες και προτείνω και την έγκριση αυτού. Όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 4, να υπενθυμίσω ότι είναι ότι ένα κονδύλι στο οποίο υπάρχουν 7,3 δις ευρώ τα οποία δεν ε, ε, απορροφήθηκαν θα δοθούν για τα κράτη-μέλη αλλά θα δημιουργήσουν προβλήματα για τις πληρωμές στο πολιτές πλαίσιο ε, τα επόμενα χρόνια και να πω επίσης ότι αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού είναι σημαντικό για να ρυθμίσουμε την κατάσταση της μετανάστευσης και υπάρχει θέμα και στο οργανώμα γραμμά της Frontex, για παράδειγμα. Για να βοηθήσουμε λοιπόν ε, και ε, στην επίλυση του προβλήματος των προσφύγων και επειδή ε, το Ταμείο Βοήθειας προς τους Πρόσφυγες στην Τουρκία είναι ένα ταμείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη χρήση κονδυλίων. Προτείνω λοιπόν να δοθούν προκαταβολικά 400 εκατομμύρια προκειμένου να διευκολύνουμε αυτό το ταμείο για τους πρόσφυγες. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια έκθεση για την κινητοποίηση αυτού του ποσού. Έχουμε στο τίτλο 2 ένα περιθώριο, μπορούμε να πάρουμε εκεί τα 400 εκατομμύρια. Και η πρόταση λοιπόν είναι ε, να ε, δοθεί αυτό γιατί θα βοηθήσει και τον προπολογισμό του 2016 και του 2017. Το 5-6-7 έχετε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Εδώ προβλέπετε για το 4 να σας δώσουμε και τις επόμενες ώρες το κείμενο και να υπενθυμίσω ότι στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6 θα προτείνω να μειώσουμε την ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι το τέλος της ε, διαπραγμάτευσης, δηλαδή στις 17 Νοεμβρίου, για να έχουμε και τα αποτελέσματα της συνδιαλλαγής ε, και να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Το 6 όμως προχωρά εκ παραλλήλου με την έκθεση της Μόνικα Χολμάιερ, επομένως η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών θα είναι Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στις 6 ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν θα προκύψει βάσει και της διαδικασίας του προπολογισμού που έχουμε εξελίξει. Παρατηρήσεις, ερωτήσεις, όχι. Ευχαριστώ πολύ το Ζωζέ Μανουέλ για αυτές τις ανακοινώσεις. Έχουμε λοιπόν αυτά τους ε, τρεις ε, διορθωτικούς προπολογισμούς. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα γιατί ε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχουμε διπλά. Ε, έχουμε τη διαδικασία του προπολογισμού και τη διαπραγμάτευση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είπαμε ότι πρέπει να δούμε την κατάσταση για τις εξελίξεις της συνδιαλλαγής στις 10.30. Είναι 10 η ώρα. Προτείνω λοιπόν να διακόψουμε τώρα και να συνεχίσουμε στις 10.30 και κλεισμένο των θυρών. Euh, Προβλεπόταν για τις 10.30 και και κάποιοι από τους συναδέλφους έχουν προβλέψει να έρθουν στις 10.30. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να διακόψουμε και να συνεχίσουμε στις 10.30.